Good morning, dear colleagues. Καλημέρα συνάδελφοι και συναδελφέ. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ελπίζω το καλοκαίρι να ήταν χρήσιμο για σας να, μπορέσατε, να έχετε μπορέσει να ξεκουραστείτε, να φορτίσετε τις μπαταρίες σας. Έχουμε πολλή δουλειά που μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσετε να ξεκουραστείτε, να περάσατε καλές καλοκαιρινές διακοπές και σας καλωσορίζω ξανά στην Επιτροπή μας. Ξεκινούμε λοιπόν με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν συμφωνείτε όλοι και όλες με την ημερήσια διάταξη δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καλώς. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο. Ε, ε, έγκριση των πρακτικών της 22ης ε, Ιουλίου. Έχετε κάποιο ερώτημα, έχετε κάποιο θέμα για την προηγούμενη συνεδρίαση. Εάν όχι, Περνούμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση προς το παρόν. Σημείο 5. Ανακοινώσεις της Προέδρου ως προς τις αποφάσεις των συντονιστών. Θα τα λάβετε όλα αυτά, όμως αυτά τα οποία ήδη πρέπει να γνωρίζουμε όλοι οι υπόλοιποι είναι τα εξής. Ως προς τις ακροάσεις που θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες εβδομάδες, τις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων, ως προς το θέμα αυτό, λοιπόν, οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν να σταλεί νέα επιστολή στον κύριο Γιούγκερ, με την οποία θα εκφράζουμε την ανησυχία μας τις ανησυχίες μας για τα νέα που φτάνουν στα αυτιά μας για τη σύνθεση του σώματος των επιτρόπων, όπου δεν θα ε, εκπληρωθεί μία προϋπόθεση, ένα θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς, η ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στη θεσμική εκπροσώπηση, δηλαδή στο σώμα των επιτρόπων. Ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα και για άλλους φορείς και για άλλα θεσμικά όργανα. Επομένως, Ήδη στείλαμε μια τέτοια επιστολή στις αρχές του καλοκαιριού και δεν ελήφθη ιδιαίτερος υπόψη. Θα πρέπει να επιμείνουμε περαιτέρω και να ασκήσουμε πίεση για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Άλλωστε, το Κοινοβούλιο είναι αυτό το φύση, θα εγκρίνει την νέα επιτροπή σε σώμα και δεν μπορούμε να θεωρούμε και να πιστεύουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που το 52% του πληθυσμού είναι γυναίκες, η εκπροσώπηση αυτών θα είναι τόσο ελάχιστη όσο φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή. Επομένως, ε, η πλειονότητα των συντονιστών των πολιτικών ομάδων εξέφρασαν τη συμφωνία τους με αυτή την πρόταση και θα αποσταλεί νέα επιστολή στον ε, νέο πρόεδρο κύριο Γιούνκερ και θα αποσταλεί και νέα επιστολή στην Ιταλική Προεδρία για την οδηγία για τη μητρότητα και θεωρούμε ότι το Συμβούλιο πρέπει να κινητοποιηθεί ως προς το θέμα αυτό. Άλλωστε έγινε συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Θέλουμε να μπούμε σε διάλογο, σε συζήτηση με το Συμβούλιο. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρξουν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό θα στείλουμε επιστολή με τέτοιο περιεχόμενο στην Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εγκρίναμε τη σύνταξη έκθεσης με εισηγητή από την ομάδα των σοσιαλιστών και με θέμα τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων από το 2015 και μετά. Στη δική μας Επιτροπή πρέπει ήδη να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε και να ε, δώσουμε σε αυτό που θα αναλάβει ως αρμοδιότητα την πολιτική για τη διάσταση του φύλου, για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσουμε λοιπόν ε, σε, στην, στον νέο επίτροπο ή, ε, ή στη νέα επίτροπο τις προτάσεις μας για να προχωρήσουν τα πράγματα. Στις 5 Μαρτίου του 2015 θα είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες και θα τη γιορτάσουμε στην Επιτροπή μας. Κατά τα λοιπά. Αν συμφωνείτε, μετά από αυτές τις ανακοινώσεις, μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία του προϋπολογισμού για το 2015. bueno, Καλώς. Εάν έχετε την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας, εάν την έχετε ετοιμάσει, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσει η ψηφοφορία λοιπόν. Και πρώτα απ' όλα να σα πω κάτι. Ορισμένοι συνάδελφοι μας μετέφεραν την ύπαρξη ορισμένων προβλημάτων και κάποιων ασαφιών στη μετάφραση σε ορισμένες γλώσσες. Ε, οι γλωσσικές εκδοχές δηλαδή ενδεχομένως παρουσιάζουν κάποιες ασάφειες. Όλοι να γνωρίζουμε ότι οριστική ε, και επίσημη εκδοχή του κειμένου είναι ε, το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Αφού λοιπόν μας το είπαν κάποιοι συνάδελφοι αυτό, να σας πω ότι η επίσημη εκδοχή του κειμένου είναι αυτή που έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και επ' αυτής ψηφίζουμε. Επίσης, πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, να σας πω ότι υπάρχει και προφορική τροπολογία, την οποία υποβάλλω εγώ ίδια. 6, 2, 4, 3. Εκεί ε, θέλουμε να προσθέσουμε. With particular attention should be given to Με ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί όπως το βλέπετε στο κείμενο. Αντιστήθεται δηλαδή αυτό στο υπάρχον κείμενο. Συμφωνείτε με όλα αυτά. Εάν ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. η πρώτη ψηφοφορία που κάνουμε στη νέα κοινοβουλευτική μας επιτροπή ή τουλάχιστον η πρώτη ψηφοφορία που κάνω εγώ ως προεδρεύουσα. Και αν υπάρξει διαδικαστικό πρόβλημα, ε, σας ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 λοιπόν, ψηφίζουμε. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η συμβιβαστική τροπολογία. Περνούμε τώρα στην τροπολογία 7201. 7201, όχι, 6201, ε, ε, συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 6202, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογ... Συμβιβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η συμβιβαστική τροπολογία 2. Τροπολογία 6204. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Εδώ θα πρέπει να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά ενδεχομένως. Άρχεται η ψηφοφορία 6204 για αυτή την τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι και όλες πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ 13 κατά. 62-05 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. «62.07 υπέρ» κατά «αποχές εγκρίνεται. 6208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6209 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε, θα το επαληθεύσουμε. 6209. Άρχεται η ψηφοφορία. Ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πέρας της ψηφοφορίας και σημειώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με μία ε, κάρτα εγκρίνεται. 18 ψήφοι υπέρ, 13 κατά. Είναι 12 που εμφανίζεται στην οθόνη, συν ε, η ηλεκτρονική κάρτα της βουλευτού που ήταν κατά. 62-35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62-42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62-10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνούμε τώρα την 6234 υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά προτιμώ να το παληθεύσουμε. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 6234. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 ψηφί, υπέρ, 20 κατά. 62-47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62-12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62-13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. στην οποία ενσωματώνεται η προφορική τροπολογία στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή της παρέμβασής μου. Και βεβαίως αν υπάρχουν αντιρρήσεις με στην προφορική τροπολογία να το πείτε. Ιδαλλιώς το ενσωματώνουμε και ψηφίζουμε αυτή την τροπολογία σε δύο τμήματα. Όχι, δεν θέλετε. Ψηφίζουμε λοιπόν την 6243. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6214 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστροποτική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 5. Περνούμε στην 6216. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6217 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6218 υπέρ κατά, αποχές, 6219 με προφορική τροπολογία που υπάρχει στο ε, το κείμενό της, στο, στο κατάλογο ψηφοφοριών, το έχετε. Αν δεν έχετε πρόβλημα με την προφορική τροπολογία, την ενσωματώνουμε στην 6219 και ψηφίζουμε την 6219. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62-20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62-21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62-22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62-23 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 62-24 υπέρ, κατά, αποχές, συγγνώμη, ας το επαληθεύσουμε δια της ηλεκτρονικής οδού, 62-24, ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται 18 υπέρ 14 κατά. 62-25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62-26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62-27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 6. Ποιος και ποια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62-38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62-29. Όχι. 62-30. 62-30 υπέρ. Κατά. Θα το επαληθεύσουμε για της ηλεκτρονικής οδού. 62-30 ψηφίζουμε τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, 14 κατά και 3 αποχές. 62-36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62-37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62-40 υπέρ κατά αποχές α, ε, απορρίπτεται 62-41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ψηφοφορία της έκθεσής μας για τον ε, προϋπολογισμό και περνάμε ψηφίσαμε τις τροπολογίες δεν έχουμε ψηφίσει την ε, τελική έκθεση Bueno, pues damos comienzo. Ξεκινούμε λοιπόν. Damos comienzo. Ξεκινάει το εργαστήριο. Παρακαλώ Eh, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το εργαστήριό μας. Παρακαλώ, ε, καθίστε και αν κάποιος από την αίθουσα ή κάποια από την αίθουσα ε, ε, θέλει να παραμείνει, ευχαρίστως να παραμείνει. Αλλιώς να υπάρξει περισσότερη ησυχία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Bueno, pues damos comienzo con, con este workshop eh, que se Ξεκινούμε λοιπόν με αυτό το εργαστήριο το οποίο η Επιτροπή μας έχει οργανώσει. Νομίζω ότι στις διάφορες επιμέρους συνεδρίες τις οποίες θα παρακολουθήσετε καταφέραμε να τις οργανώσουμε έτσι ώστε να τεθούν τα πιο βασικά και πιο σημαντικά θέματα. Αυτά θα μας χρησιμεύσουν θα μας χρησιμεύσουν για να κάνουμε μια επισκόπηση των πιο φλεγόντων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φύλων. Ε, τα πιο σημαντικά λοιπόν τα έχουμε θέσει ως θέματα συζήτησης στις διαφορετικές συνεδρίες. Παρακαλώ, είναι πολύ δύσκολο να προεδρεύσω και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλούμε και να προχωρούμε με τόσους πολλούς ανθρώπους σε αυτή την αίθουσα και μάλιστα ορθίους. Eh, Ελπίζω λοιπόν να μπορέσω να ε, συνεχίσω. Ε, λοιπόν, έλεγα ότι Έχουμε έξι διαφορετικά τμήματα, ε, έτσι έχουμε χωρίσει αυτό το εργαστήριο και σε κάθε τμήμα ε, προσπαθούμε να ασχοληθούμε με ένα από τα πιο σημαντικά θέματα ε, για την ισότητα των φύλων. Θέμα το οποίο την χάνει επεξεργασία σε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Και πάντοτε εν ώψη της νέας στρατηγικής μετά το 2015. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η δική μας Επιτροπή μπορεί να συμβάλλει στο έργο που θα γίνει τους επόμενους επόμενους μήνες και ε, περισσότερο βεβαίως. Καταρχάς, να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς που θα συμμετάσχουν, ε, όλους και όλες αυτές που θα μοιραστούν μαζί μας ε, τις γνώσεις τους για τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή επιτάπητος. Έχουμε λίγο καθυστερήσει. Ξεκινούμε με το πρώτο gender mainstreaming, budgeting και monitoring, η ισότητα των φύλων, η ένταξη του, της διάστασης του φύλου και στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό, για όλες τις υπόλοιπες πολιτικές και το monitoring, η παρακολούθηση. Όλα αυτά, εποπτεία, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Η καθηγήτρια κυρία Φιώνα Μπέβεριτς, από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ θα πάρει το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι για μένα μεγάλη τιμή η παρουσία μου εδώ σε αυτή το εργαστήριό σας. Στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ με συνοδεύει και η κυρία Ζέντζικ καθώς και η κυρία Ντράιγουντ από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. Θα καλύψω το θέμα της ισότητας των φύλων, των προϋπολογισμών για την καταπολέμηση της ανισότητας και την εποπτεία. Τις συστάσεις και τα συμπεράσματα τα βλέπετε στις σελίδες 25 και 26. Σήμερα όμως στην παρουσίασή μου θα περιοριστώ στη σύνοψη σελίδες 9 με 10. Με 10. Όχι, δεν έχει. Δεν. Οικονομία. Όπως ξέρετε η στρατηγική για την ισότητα των φύλων βασίζεται σε δύο στοιχεία την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς και πρώτα και μετά συγκεκριμένα μέτρα. Η γενική στρατηγική μας δίνει την ευκαιρία να δούμε αν αυτή η βασική αρχιτεκτονική δυτή παραμένει βιώσιμη και σωστή. Βρίσκουμε ότι ναι. Γιατί υπάρχουν πολλά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πολύπλοκο πρόβλημα της ανισότητας των φύλων. Γενικά θεωρούμε ότι τα προβλήματα των φύλων μπορούν να, να αντιμετωπιστούν από ενωσιακή πολιτική εφόσον υπάρξει πολιτική θέληση. Η Ένωση πρέπει να αναμειγνύει εθελοντικά και υποχρεωτικά μέτρα δεσμευτικά αν και η νομοθετική δράση της δεν ήταν και τόσο συνεπής τα τελευταία χρόνια από το 10 και μετά αλλά παραμένει ένα βασικό εργαλείο. Τα δεσμευτικά μέτρα σε συγκεκριμένους τομείς διασφαλίζουν ότι θα υπάρχουν σαφείς κανόνες και προσδοκίες έτσι ώστε η Ένωση να μπορεί να συνεχίσει να καθορίζει τα ελάχιστα τουλάχιστον κριτήρια ώστε να υπάρχει ισοτιμία στους κανόνες μεταξύ ας πούμε των προμηθευτών υπηρεσιών και των εργοδοτών. Ένα παράδειγμα της χρήσης των δεσμευτικών μέτρων υπέρ της ισότητας των φύλων είναι ο κανονισμός, ή κανόνες μάλλον για την ισότητα των φύλων που προβλέπει το πρόγραμμα Horizon 2020. για την ισότητα των φύλων σε τομείς όπου δεν υπήρξε και μεγάλη πρόοδος. Ιδιαίτερα οι κανόνες αυτοί ε, είναι υποχρεωτικοί για όλα τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι και τα λεγόμενα soft μαλακά μέτρα και τα δεσμευτικά είναι χρήσιμα. Γι' αυτό υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει αυτή η διπλή αντιμετώπιση για την επίλυση του προβλήματος και αυτό δεν έχει αλλάξει στη νέα στρατηγική. Η στρατηγική 10 με 15 προέβλεπε πέντε τομεί προτεραιότητας και οι αιτήσει εκθέσει δείχνουν ότι έχει συμβεί κάποια, έχει μειωθεί κάποια πρόοδο σε μερικού τομεί, αλλά α, όχι ομοιόμορφα. Η έγκριση μιας νέας στρατηγικής μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε πού ακριβώς έχει σημειωθεί η πρόοδος και πόση και ποια είναι τα κυριό, ποιοι είναι οι κυριότεροι τομείς που πρέπει να, στους οποίους πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Μας δίνει επίσης την ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τις ε, υποστηρικτικές στρατηγικές για να δούμε πώς θα μπορούσαν να σημειωθούν βελτιώσεις και, και στα όργανα της Ένωσης και στα κράτη-μέλη. Μπορούμε να σημειώσουμε ότι το Συμβούλιο ήδη ζήτησε από τα κράτη-μέλη το Δεκέμβριο του 2013 να διατηρήσουν την επιβολή κρατικών μέτρων για την ισότητα των φύλων γενικά για την Ένωση Πρόκειται για εξέλιξη, μάλλον παρά για επανάσταση στη στρατηγική αυτή, με βάση ό,τι μάθαμε από την προηγούμενη στρατηγική. Λοιπόν, η εποπτεία, η επιτήρηση της εφαρμογή της πολιτικής για την ισότητα των φύλων είναι κάτι βασικό, αν και είναι πολύπλοκο πρόβλημα. Η στρατηγική ισότητα των φύλων δείχνει ότι δεν είναι εύκολο να σημειώσουμε, να δούμε πού ακριβώς υπήρξε πρόοδος και πού η παναχώρηση. Γι' αυτό η εποπτεία είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Από τότε που εγκρίθηκε η προηγούμενη στρατηγική βελτιώθηκε η δυνατότητα της Ένωσης να γνωρίζει πώς έχουν τα πράγματα μέσω του καθορισμού της Υπηρεσίας για την Ισότητα των Φύλων, του Οργανισμού για την Ισότητα των Φύλων. Ήδη οι μελέτες που έχουν συγκράψει από το, την ίδρυσή τους δείχνουν ότι οι δυνατότητες τεχνογνώσης και πληροφόρησης του οργανισμού αυτού είναι σημαντικές. Θεωρούμε λοιπόν ότι στη νέα στρατηγική πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο οργανισμός αυτός για να μπορεί να ταυτίζει πού βρίσκονται τα προβλήματα και πώς μπορούν να βρεθούν οι λύσεις. Είναι ένας νέος πόρος λοιπόν στη στρατηγική αυτή ισότητα των φύλων για περισσότερη αποτελεσματικότητα. Η πραγματική αποτελεσματική εποπτεία σημαίνει ότι πρέπει να δούμε και αν υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις ή χάσματα στην πληροφόρησή μας. Ο δείκτης της ισότητας των φύλων είναι κάτι που μας επιτρέπει να σημειώσουμε ακριβώς τις πρόοδους, να διαπιστώσουμε. Για τη βία μεταξύ των φύλων ακόμα συζητιέται το ποιο θα μπορούσε να είναι το καλύτερο εργαλείο αντιμετώπισης και οι εμπειρογνώμονες και οι πολιτικοί συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να βρεθεί ένας τρόπος να έχουμε στοιχεία και για αυτό το θέμα. Η νέα λοιπόν στρατηγική πρέπει να μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα καθορίζοντας ας πούμε συγκεκριμένους στόχους και κλίμακες. Ο δείκτης αυτός που άρχισε να εφαρμόζει από το 13 το ΆΙΓΕ, το Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων, θα επιτρέψει την επιτήρηση, των, την υποπτία των δεδομένων αυτών για ολόκληρη την Ένωση. Είναι εργαλείο πολύ πλήρες και συστήνουμε ο δίκτυς αυτός να συμπεριλαμβάνεται στη νέα στρατηγική ως μηχανισμός εποπτείας και τα κράτη-μέλη καθώς και η Ένωση καθεαυτήν να θέσουν ορισμένους συγκεκριμένους στόχους για τη βελτίωση του θέματος της ισότητας των φύλων με βάση τα στοιχεία του δείκτη αυτού. Η επιμόρφωση των φύλων τώρα για τα φύλλα, για την ισότητα Στην προσθήκη 3 της εκθεσής μας το αναφέρουμε αυτό συγκεκριμένα γιατί δεν είναι πολύ εύκολο και εδώ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Συστήνουμε λοιπόν στις χώρες μέλη και την Κομισιόν να δοθεί περισσότερη προσοχή στο θέμα αυτό του gender training ώστε να διασφαλίζονται οι δεξιότητες και των δύο φύλων για την καλύτερη δυνατή χρήση. Επίσης η αξιολόγηση της πολιτικής για την ισότητα των φύλων. Υπάρχουν συγκεκριμένες αδυναμίες στο πλαίσιο αξιολόγηση που κάνει γι' αυτό το θέμα η Ένωση ως προς τα ε, φύλλα. Και ιδιαίτερα η Κομισιόν θα μπορούσε να επωφεληθεί περισσότερο από ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Επίσης, θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο τα κράτη-μέλη να κάνουν τις αξιολογήσεις αυτές, γιατί μερικά έχουν μεγάλες ελλείψεις. Τώρα τα στερεότυπα για τα φύλλα. Αυτά η ύπαρξή τους υπονομεύει την οικονομική και στρατηγική και τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων και πρέπει κάτι να γίνει. Είναι και αυτό κάτι πολύπλοκο γιατί οι κύριες δικαιοδοσίες ευθύνε είναι των κρατών μελών και φυσικά υπάρχουν εδώ τίθενται θέματα και ελεύθερης έκφρασης, ελευθερίας έκφρασης. Υπάρχουν όμως επιχειρήματα υπέρ της λήψης ορισμένων συγκεκριμένων ενωσιακών μέτρων. Παραδείγματος χάρη μερικά χώρες μέλη είναι διατεθειμένες να καταπολεμήσουν πιο στεναρά την σεξιστική διαφήμιση εφόσον αυτό δεν διαταράξει την ενιαία αγορά. Η σύστασή μας είναι να οργανωθεί μια μελέτη για το θέμα αυτό και υποστηρίζουμε τη σύσταση για, της Επιτροπής για, από το 2010 να υπάρξει επιτέλους ένας κοινός ορισμός για το τι είναι σεξιστικές εικόνες και στερεότυπα. Και τέλος, οι προϋπολογισμοί για όλα αυτά gender budgeting. Εδώ τα κράτη-μέλη και τα διεθνή ήθη έχουν προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια γιατί τώρα γίνεται κατανοητό ότι και οι προλογισμοί ακόμα δεν είναι ουδέτεροι ως προς τα φύλλα. Οι δημοσιονομικοί στόχοι λοιπόν πρέπει να εξεταστούν και από απόψεως φύλων έτσι ώστε να ταυτιστούν πρώτα τα προβλήματα και μετά να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε οι δαπάνες σε έναν τομέα να μην ακυρώνονται από την έλλειψη πόρων σε άλλο τομέα. Όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται και για μια ευκαιρία οι διαδικασίες έγκρισης προϋπολογισμών και δαπανών να είναι και πιο υπόλογες στους επόπτες. Γι' αυτό συστήνουμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με τη στήριξη της Κομισιόν να θέσουν τέτοιο θέμα ισότητας φίλων και στον προϋπολογισμό. Τον ενωσιακό προϋπολογισμό και το ΠολΔΙΠ, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρόσφατα το Συμβούλιο ζήτησε να προσθεθεί ένας πυλώνας φύλων στη γενική οικονομική μας στρατηγική. Και τέλος, σε εποχές δημοσιονομικής κρίσης φαίνεται ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει ως προς τα φύλλα και την κρίση συστήνουμε να υπάρξει συστηματική εξέταση της κατάστασης που αφορά τα φύλλα και σε περιόδους κρίσης όπως και στις υπόλοιπες περιόδους. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε καθηγητά, καθηγήτρια Μπέβεριτζ. Τώρα υπάρχει δυνατότητα οι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο για ερωτήσεις αλλά και για απαντήσεις. 20 λεπτά. Ποιος θέλει να θέσει ερώτημα. Εγώ είμαι από την Ουγγαρία, είμαι ευρωβουλευτής από την Ουγγαρία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζονται πολλά, προφανώς και στη δική μου τη χώρα. Έχουμε πολλούς ε, ανθρώπους, πολλές γυναίκες και πολλά παιδιά που ζουν σε άθλιες ε, συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν εμένα δεν μου αρέσει να γίνεται ε, γενικά λόγος για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί υπάρχουν ε, δυστυχώς ε, χώρες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας ε, στο βορρά και αντίστοιχα στο νότο της Ευρώπης. Υπάρχουν πολύ λίγοι που επισκέπτονται σκέπτονται τι συνεδριάση μας και θέλω να σας παρακαλέσω όσοι εδώ ενοχλούν και θέλουν να πιούν καφέ με κάποιον άλλον να τους παρακαλέσετε κύριε Πρόεδρε να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Μπορούμε να ε, συγκεντρωθούμε καλύτερα στη δουλειά μας. Μιλάμε λοιπόν για άντρες ή για γυναίκες που είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τις ε, οικογένειές τους και να μεταβούν σε πιο πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπηρετήσουν τις χώρες αυτές, ε, εργάζονται σε άθλιες συνθήκες, ε, ε, μη ελεγχόμενες, εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί. Τελικά υπάρχουν και πολλοί που δυστυχώς καταλήγουν θύματα του, της εμπορίας ανθρώπων. Ε, υπάρχουν γυναίκες που εκπορνεύονται. Πώς είναι, δυνατόν, πώς είναι λοιπόν δυνατόν να μιλάμε για μια ενιαία Ευρώπη τη στιγμή που υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, σε αυτή την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά βέβαια, ενώ έχουμε πολλές ε, γυναίκες οι οποίες όπως σας είπα ζουν στην απόλυτη εξατλίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη πριν από μισή ώρα υπερψηφίσαμε τεράστια κονδύλια για εκπαίδευση, για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε διάφορες πολιτικές. Για όλα αυτά εγκρίθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και θέλω να ρωτήσω, οι γυναίκες της Ανατολικής Ευρώπης σε τι θα επωφεληθούν από όλα αυτά. Μιλάμε για γυναίκες οι οποίες σας είπα ζουν σε απόλυτη εξαθλίωση. Μήπως μπορείτε με λίγα λόγια να μας πείτε όλα αυτά τα τεράστια κονδύλια τα οποία προβλέφτηκαν κατά τα τελευταία χρόνια στους ενωσιακούς προϋπολογισμούς, αυτά τα χρήματα πώς ακριβώς βελτίωσαν την καθημερινότητα των γυναικών στις μετακομμουνιστικές χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την απάντησή σας. I, I think this is, um, Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα που δείχνει με απόλυτη σαφήνεια τη σημασία της ένταξης της διάστασης του φύλου σε διάφορες πολιτικές. Υπάρχουν οι πολιτικές του Κοινωνικού Ταμείου, του Περιφερειακού Ταμείου, όπου όπως είπατε εκταμιεύονται πολύ ψηλά κονδύλια για διάφορες πρωτοβουλίες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε τα θέματα της ισότητας των δύο φίλων σε διάφορες ε, πολιτικές. Ε, όσον αφορά τώρα την ένταξη της ε, διάστασης του φίλου, θα πρέπει να ελέγχουμε τι ακριβώς γίνεται όταν εκταμιεύονται, όπως σας είπα, τα κονδύλια να ελέγχουμε ποιες είναι ακριβώς οι επιπτώσεις σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών Ακριβώς αυτό θέλω και εγώ να πω, ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος, χρειαζόμαστε τη διαφάνεια. Πρέπει να κατανοήσουμε επακριβώς ε, τις ε, επιπτώσεις σε άνδρες, γυναίκες και σε άλλες ομάδες της κοινωνίας. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μειονεκτούσες ομάδες. Uh, uh, και επίση ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, σε μειονεκτική θέση όσον αφορά όλα αυτά τα οποία προανέφερα. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερος για την παρουσίαση αυτή. Θα ήθελα να ρωτήσω την καθηγήτρια κυρία Μπέβεριτς το εξής. Προλίγου στην Ισπανία, αλλά ούτως ή άλλως αυτό έχει υποθεί και στην Ευρωστάτα, ε, ζητήθηκε στον υπολογισμό του Εθνικού ΑΕΠ να ε, λαμβάνεται υπόψη ε, ένα ζήτημα ή μάλλον πολλά ζητήματα τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα. Π.χ. Ε, το προϊόν το οικονομικό από την πορνεία, δηλαδή το οικονομικό όφελος που προκύπτει η συναλλαγή ε, να ενσωματώνεται στον τρόπο υπολογισμού του ΑΕΠ μιας χώρας. Και την άλλη εκτιλήσεται η συζήτηση για την νομιμοποίηση ή μη νομιμοποίηση της πορνείας. Όλα αυτά είχαν τεράστια αντίκτυπο στη κοινή γνώμη. Επομένως, ε, το να ληφθεί η διάσταση του φύλου υπόψη στον προϋπολογισμό και στα οικονομικά ε, σημαίνει ότι θα λάβουμε υπόψη μας ε, και το οικονομικό όφελος που δημιουργείται από την πορνεία και από την συναλλαγή. Το να θέλουμε gender budgeting σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχόμαστε κάτι τέτοιο και αν ναι, κατά τη γνώμη μου αυτό είναι κάτι το αρνητικό. Από εκεί και πέρα. θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο η δημόσια διοίκηση ε, στην οποία αναφερθήκατε ε, θα πρέπει να πορευτεί. Ε, πολύ συχνά διαφάνεια σημαίνει, είναι, ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει ένα ευρώ για κάποιον ο οποίος το, το δαπανά για χύψη λόγο. Αλλά δεν γίνεται σχεδόν ποτέ αξιολόγηση του οικονομικού αποτελέσματος, του αποτελέσματος ε, ε, που προέκυψε από τη δαπάνη. Δεν γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου, του κινδύνου ε, να χάσουμε ή να μην αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια ή τελικά να μην φέρουν καρπούς, αλλά ο κίνδυνος αξίζει τον κόπο εάν καταφέρουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αυτό, γι' αυτό δεν, δεν συζητούμε πολύ. Θα πρέπει να έχουμε λογιστικά αποτελέσματα αλλά να έχουμε και πολιτικές αποφάσεις και για να πάρθει πολιτική απόφαση συχνά θα πρέπει να αναλαμβάνεται και ο αντίστοιχος κίνδυνος κατά τη γνώμη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για το budgeting του, ε, σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και όπως σας είπα, Υπάρχουν κάποιε καλέ πρακτικέ. Βεβαίω υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά για να αποδείξουμε ότι αυτό είναι ένα αποτελεσματικό μηχανισμό. Όμω Τώρα πλέον έχει γίνει κατανοητό το όλο θέμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει πώς μπορεί ορισμένα στοιχεία της, ε, της ισότητας των δύο φύλων να τα εντάξει στους προϋπολογισμούς της. Κοιτάξτε, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι οποτεδήποτε δαπανώνται χρήματα για ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί να υπάρξουν συγκεκριμένες επιπτώσεις σε μια συγκεκριμένη ομάδα γυναικών σε κάποια κρατημέλη όπως αναφέρθηκε αλλά πράγματι τα χρήματα δεν φτάνουν εκεί που θα έπρεπε. το budgeting, η ένταξη της διάστασης του φύλου στον προπολογισμό είναι μια ευκαιρία για να ε, εντοπίσουμε ακριβώς για πόσα χρήματα μιλάμε και για να έχουμε μια ευκαιρία να ελέγξουμε κατά πόσον ο στόχος επιτεύχθηκε ή όχι. Και αν όχι, ε, ποια ακριβώς ήταν τα εμπόδια που παρεμπόδισαν μια απόφαση υψηλού επίπεδου να φτάσει στην φάση ε, ενώ πολλοί από αυτούς που έλαβαν τις αποφάσεις είχαν θεωρήσει ότι ε, πράγματι αυτό ε, θα έφτανε στην καθημερινότητα. Βλέπουμε ότι οι αποφάσεις υψηλού επίπεδου βασίζονται σε κάποιες παραδοχές, αλλά δυστυχώς πολύ συχνά δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των δαπανών μέχρι που να φτάσουν στον τελικό αποδέκτη. Και πιστεύουμε ότι υπήρξαν επιπτώσεις που όμως δεν υπήρξαν. Το gender budgeting λοιπόν είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε, όπως σας είπα, να εξετάζουμε τις συγκεκριμένες συνέπειες ε, σε συγκεκριμένες ομάδες για να δούμε αν πραγματικά υπήρξαν τα εκτέ ε, αποτελέσματα. Ε, δυστυχώς, ε, ναι, αν έχετε καλώς το μικρόφωνο. Για την πρώτη ερώτηση που σας έκανα, από τη στιγμή που εσείς είστε επιρρογνώμονα στο θέμα του gender budgeting, ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την πρόταση η ίδια τα γη της Ευρωστάτ. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η Ισπανική κυβέρνηση δεν θέλησε να κάνει κάτι άλλο. Η Ευρωστάτ διέταξε να εντάσσεται ως λογιστική εγγραφή στο εθνικό ΑΕΠ, δηλαδή με θετικό πρόσημο στο ενεργητικό, ε, το ε, οικονομικό προϊόν από την ε, από τις συναλλαγές της πορνείας. Η Ευρωστάτα παρουσιάζει στατιστικές θεωρούν ότι ε, αυτά τα οικονομικά νούμερα είναι υπέρ του πλούτου της χώρας. Ποια είναι η γνώμη σας. Δεν είμαι οικονομολόγος και δεν θέλω να τοποθετηθώ πολύ σε αυτή την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την έννοια ότι δεν μιλάμε μόνο για τα έσοδα από την πορνεία, αλλά και από πολλές άλλες δραστηριότητες που ε, δεν καταγράφονται. Τώρα, κατά πόσον αυτό σημαίνει ε, ή ότι υπάρχουν κάποιοι που επωφελούνται και άλλοι υποφέρουν από αυτές τις συναλλαγές ε, Τόντι δεν, είναι, δεν επικρατεί διάβια. Υπάρχει η αδιαφανής αλλά και η διαφανής οικονομία και πρέπει να τα εξετάσουμε. Ε, μιλάμε όμως ε, για ένα πολύ δύσκολο θέμα που υφίσταται εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι απλά ένα θέμα που αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Είναι ένα τεράστιο θέμα που αφορά, όπως σας είπα, την αδιαφάνεια της οικονομίας. Και επειδή όμως δεν είμαι οικονομολόγος, επιτρέψτε μου να σταματήσω εδώ. Σας ε, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπεβερέτς. Εάν λοιπόν ε, δεν υπάρχουν άλλες ε, ερωτήσεις επί του θέματος, θα συνεχίσουμε το εργαστήριό μας και η επόμενη εμπειρογνώμονας θα αναφερθεί στην οικονομική ανεξαρτησία και στη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Μαρτσέλα Κόρση από το Πανεπιστήμιο Λασαπιέντσα της Ρώμης να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να σας απευθύνω σήμερα το λόγο. Ε, βρισκόμαστε στην αρχή ε, μιας ε, νέας κοινοβουλευτικής θητείας που συμπίπτει και γενικότερα με νέες θεσμικές εξελίξεις. Η δική μου λοιπόν η δουλειά νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολη γιατί δεν έχω αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου και εγώ λοιπόν θα αναφερθώ στο έγγραφο το οποίο διανεμήθηκε σήμερα και ξεκινάει με τη σελίδα 38 και ε, όπου θα αναφέρομαι και θα παραπέμπω σε γραφήματα θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω ε, να ανατρέχετε στις διαφάνειες μιλάμε για τη δική μου νομιλία που είναι από τη σελίδα 57 και ό,τι ακολουθεί περαιτέρω. Απλά αυτό για να παρακολουθείτε λιγάκι αυτά που θα σας πω, τις πληροφορίες που θα αναφέρω. Μιλάμε λοιπόν για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και κυρίως μιλάμε για το ρόλο που διαδραματίζουν στην αγορά εργασίας. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ε, έχει εξεταστεί ε, επανειλημμένα ε, και εγώ δεν είμαι οικονομολόγος όπως και η συνάδελφός μου, όμως θα Ήθελα να σας δώσω ένα πιο καθαρό παράδειγμα και θέλησα λοιπόν τη δική μου την έκθεση να τη βασίσω σε, ορισμένα, σε συγκεκριμένα στοιχεία στα οποία θα αναφερθώ και ευθύ αμέσω. Βεβαίως ε, θα πρέπει να ξεκινήσω από κάτι το οποίο γνωρίζουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα θέματα που συζητάμε και μερικοί εξημών εξάλλου έχουν και θεσμικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτά τα θέματα. Να πω λοιπόν το εξή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που διονύζεται, πρόκειται για την περιθωριοποίηση της γυναίκας ε, που εργάζεται στις αγορές εργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, κάποιες αλλαγές, αλλά παρόλα αυτά το γεγονός αυτό εξακολουθεί να υφίσταται. Περιφερειοποίηση λοιπόν με διάφορες μορφές και μία από τις σημαντικότερες ε, είναι ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση των γυναικών σε ορισμένου παραγωγικούς τομείς οι οποίοι τομείς αυτής ε, παρουσιάζουν και χαρακτηρίζονται από χαμηλότερους μισθούς. Αναφέρθηκε από τη συνάδελφο από την Ουγγαρία ότι υπάρχουν περιπτώσεις πραγματικά τραγικές ε, και σε εμά στην Ιταλία ισχύει αυτό. Σε εμά στην Ιταλία υπάρχουν οι οικιακές βοηθοί που έρχονται από αυτές τις χώρες οποίες αναφέρθηκε συνάδελφος. Έχουμε λοιπόν χαμηλούς μισθούς και δυστυχώς βλέπουμε επίσης ότι στα υψηλά αξιώματα και εκεί υπάρχουν όλο και περισσότερες γυναίκες. Και αυτό επιδεινώνεται λόγω της ε, όξυνσης της κρίσης. Το τελευταίο θέμα που θα αναφερθώ είναι το θέμα των ε, συντάξεων για τις γυναίκες και ε, θα θελήσω να καλύψω και αυτό το θέμα. Όλα αυτά λοιπόν, όπως αναφέρθηκε ήδη, έχει εξεταστεί, όλο το θέμα έχει εξεταστεί από το Ινστιτούτο Ισότητας ε, των Δύο Φύλων. Υπάρχει ένας ε, δείκτης για την ισότητα των δύο φύλων και μπορείτε εδώ να δείτε τον πίνακα υπαριθμών 1 και ο πίνακας αυτός είναι μια συνθετική απαρίθμηση για την ισότητα που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλλα και βλέπουμε ότι ποικίλει από το 0 μέχρι το 100 ο δείκτης αυτός ο δείκτης, ε, όπως βλέπετε, δίνει μια συλλογική εικόνα. Και φτάνουμε στο 54. Στο 54 είναι ο μέσος όρος. Αυτό όμως ε, είναι ένα είδος εισαγωγής, απλά έτσι το αναφέρω ενδεικτικά. Και αν δούμε λιγάκι το τι καλύπτει αυτός ο δείκτης, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την εισήγηση, στα δύο θέματα που αναφέρομαι, δηλαδή στην ε, θέση απασχόλησης και στα εισοδήματα, βλέπετε ότι η κατάσταση την οποία παρουσιάζω εγώ είναι λιγάκι καλύτερη από αυτή που παρουσιάζει ο δείκτης. Βλέπουμε ε, όμως ότι υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Ε, τουλάχιστον σε αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα της δικής μου της εισήγησης. Και αυτά σας τα λέω απλά για να έχετε κατά νου κάποια συμπεράσματα που νομίζω ότι μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις αξιολογήσεις τις οποίες θα καταλήξω σήμερα και εγώ και οι συνάδελφοί μου. Αυτή λοιπόν, ε, αυτό το συμπέρασμα δεν μπορεί κανένα να το εξάγει χωρίς να ε, αγνώντας ε, την κρίση, χωρίς να λάβει υπόψη του τη επιπτώσεις της κρίσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί θεσμοί, εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι, οι οποίοι έχουν εξετάσει τις επιπτώσεις της κρίσης. Ας δούμε λοιπόν η κρίση αυτή τη στιγμή ε, σε τι οδηγεί. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα δηλαδή μιλάμε ε, για μια αρχική εκτίμηση αυτή την οποία αναφέρουμε. Με την πρώτη ματιά το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι η κρίση δίνει κάποια δείγματα περίεργα, οξύμορα, αλλά αν θέλετε και επικίνδυνα σε κάποιο βαθμό. Γιατί η κρίση αρχίζει να περιορίζει το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Αυτή λοιπόν την εξέλιξη θα μπορούσε κανείς να την εκλάβει θετικά. Όμως δεν είναι, και το λέω ξεκάθαρα, το θέμα είναι ότι απλώς όλοι πάμε προς τα κάτω. Πάνε και άνδρες προς τα κάτω. Είμαστε όλοι σε χειρότερη θέση. Αυτό λοιπόν προφανώς μειώνει, οδηγεί σε μείωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων. Άρα δηλαδή η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη από αυτήν που θα σας παρουσιάσω σήμερα, όμως ε, στην έκθεση μου μπορείτε να τρέξετε και εκεί υπάρχουν και άλλα στοιχεία βιβλιογραφίας για να εμβαθύνετε, να εντρυφήσετε περισσότερο στο θέμα. Η κατάσταση λοιπόν, όπως σας είπα, ε, που παρουσιάζεται είναι ότι μειώνεται το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα, όμως επαναλαμβάνω αυτό οφείλεται στο ότι όλοι μας είμαστε σε χειρότερη κατάσταση και θα ήθελα εδώ να σας παρουσιάσω παρουσιάσω δύο γραφήματα που δείχνουν τους βασικούς δείκτες της αγοράς εργασίας. Από τη μια έχουμε το δείκτη συμμετοχής, το δείκτη ε, επαγγελματικής απασχόλησης και εκεί βλέπετε ότι υπάρχει μία ελαφρά μείωση ε, στο χάσμα των δύο φύλων από το 2006 ως το 2013. Η μείωση αυτή αφορά περισσότερο το ποσοστό απασχόλησης που όπως ξέρετε είναι ο βασικός δείκτης ε, σε σχέση με την στρατηγική του 2020. Και εκεί λοιπόν ε, το ποσοστό απασχόλησης από τη Eurostat, από ό,τι προκύπτει από τα στοιχεία της, από το 6 μέχρι το 13, εκεί υπάρχει μια σύγκληση των δύο φύλων. Γιατί, διότι το ποσοστό απασχόληση των ανδρών απλά επιδεινώνεται. Από την άλλη βέβαια βλέπουμε ότι όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, βλέπετε ε, ποιο ήταν το χάσμα στην αρχή. Οι γυναίκες ε, μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας ε, αλλά τώρα πια είναι και πολύ περισσότεροι άνεργοι άντρες. Στην, στην Αμερική γίνεται λόγος για μια ανδρική κρίση, κρίση που αφορά τους άντρες τουλάχιστον όταν ξέσπασε η κρίση. Και από ό,τι φαίνεται όμως, σιγά σιγά η κρίση αυτή έχει επεκταθεί και στις γυναίκες, γιατί πλέον η κρίση δεν έχει πλήξει μόνο τους άντρες, τους ε, κλασικά ανδρικούς ε, τομείς, αλλά η κρίση πλέον επεκτείνεται και ε, σε τομείς όπως είναι η παροχή υπηρεσιών και εκεί έχουμε πλειοψηφία γυναικών. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία δύο τρίμηνα υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία και πάλι η ανεργία των ε, γυναικών είναι μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. Πρέπει όμως και αυτό να το παρακολουθήσουμε ε, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να είμαστε σίγουροι στα συμπεράσματά μας ότι ε, πράγματι η κρίση θα πλήξει περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες κατά τους επόμενους μήνες. Και εφόσον εξάγουμε αυτά τα συμπεράσματα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και στην πολιτική που οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι και η ποιότητα της εργασίας επιδεινώνεται. Αυτό παρουσιάστηκε θαυμάσια από την έκθεση της Eurofound, ε, επιδείνωση λοιπόν της ποιότητας ε, και σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών. Βεβαίως εγώ τώρα μιλάω για τη δική μου τη χώρα, την Ιταλία. Υπάρχει μια πολύ καλή έκθεση του Ινστιτούτου ISFOL, μεταρχικά ISFOL, όπου αποδεικνύεται ότι για τρίτη φορά ε, διαπιστώνεται επιδείνωση της ποιότητας εργασίας. Γιατί συμβαίνει αυτό, διότι όλο και περισσότερο επιδεινώνονται οι συνθήκες εργασίας. Δηλαδή γίνεται όλο και περισσότερη αναφορά σε μερική απασχόληση. Ε, αυτή βέβαια είναι μια εναλλακτική λύση για την ε, μία απόλυση. Οι ίδιοι εργαζόμενοι συμμετέχουν ε, εθελοντικά σε μερική απασχόληση και εκεί προφανώς αυτό ευνοεί τις γυναίκες. Όπως σας λέω πρόκειται για μία μερική απασχόληση ε, εθελοντική αλλά και πολλές φορές μη εθελοντική. Αυτό αφορά κυρίως ε, τις νεότερες ε, γυναίκες. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στο να προσθέτει μια γύρανση του πληθυσμού και να υπάρχει και μια αναβολή της απόκτησης παιδιών, τουλάχιστον για το πρώτο παιδί. Σας λέω λοιπόν ότι η επιδείνωση των συνθηκών εργασία αφορά τις νεότερες γυναίκες. Και αν δείτε τώρα τα στοιχεία και μπορώ να σας ε, τα δείξω αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε όμως να τα δείτε και καλύτερα μόνοι σας ε, γιατί φοβάμαι ότι η δική μου διαφάνεια δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη, δεν είναι τόσο ευκρινής. Βλέπετε και εκεί λοιπόν έχω υπεριστεί το χάσμα των ε, δύο φύλων. Κάτι άλλο που αφορά στην ποιότητα εργασία είναι η εποχική εργασία, η επισφαλής θέση απασχόλησης. Τουλάχιστον στη δική μου τη χώρα αυτό είναι πλέον μια ενδυμική κατάσταση ε, είναι κάτι που υφίσταται. Για άλλη μια φορά λοιπόν θέλω να επαναλάβω, έχουμε τις άτυπες ε, συνθήκες απασχόλησης, έχουμε ε, συνθήκες ε, εργασίας που αφορούν ιδιαίτερα τους νέους και ιδιαίτερα τις νέες γυναίκες. Αυτή η εξέλιξη είναι μόνη δυνατότητα για να μπει κανεί στην αγορά εργασίας. Αυτές λοιπόν οι συμβάσεις είναι συμβάσει οι οποίε δυστυχώ σιγά σιγά νομοθετούνται κιόλα, καταχειρώνονται με νομοθετικά μέτρα. Αυτό δεν θέλω τώρα να το εξετάσω σήμερα. Βέβαια αυτό αφορά περισσότερο τι γυναίκε, περισσότερο από ότι του άντρε. Και επαναλαμβάνω ότι αυτές οι εξελίξεις καταλήγουν να είναι ενδυμική εξέλιξη κυρίως για τους νέους. Αυτά είναι τα γραφήματα στα οποία αναφέρθηκα, αλλά και πάλι σας λέω μπορείτε να τα δείτε τα γραφήματα αυτά με μεγαλύτερη προσοχή ε, στις, ε, στα έντυπα που σας διανεμήθηκαν, γιατί δεν φαίνονται καλά, δεν είναι ευκρινή αυτά τα γραφήματα τα δικά μου. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα που ήθελα να φέρω. Ο πρώτος ε, στόχος της ομιλίας μου που όπως σας είπα αυτά σας τα είπα γιατί και μου ζητήθηκα να τα πω. Ε, το πώς δηλαδή επηρεάζει η κρίση την αγορά εργασίας και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που πρέπει να εξτάσουμε και εν μέρη και αυτό έχει σχέση με τους δείκτες που σας παρουσίασα στην αρχή. Ένα άλλο θέμα είναι οι μισθολογικές διαφορές όσον αφορά τα δύο φύλλα. Ένα θέμα που έχει εξεταστεί αρκετά σε ενωσιακό επίπεδο. Η Κομισιόν ασχολήθηκε μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το αποτέλεσμα είναι ότι εκεί παρουσιάζεται μία στασιμότητα. Δεν παρουσιάζεται βελτίωση στις μισθολογικές διαφορές. Αν δείτε λιγάκι το γράφημα και νομίζω αυτό μπορείτε να το διαβάσετε καλύτερα και σας το συστήνω επιφύλακτα. Το 2008 και το 2009 βλέπετε από τότε δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές. Το τελευταίο στοιχείο που βλέπουμε είναι το 16-17% διαφορές. Ε, βεβαίως υπάρχει εδώ μια καθυστέρηση στα στοιχεία. Ε, αυτά αφορούν το 2012. Και αυτό το 16-17% είναι κατ' ουσίαν σημαίνει στασιμότητα. Τώρα ε, είμαστε σχεδόν κατά την πέμπτη χρονιά της βαθιάς κρίσης. Παρ' όλα αυτά όμως ε, οι δείκτες αυτής της μορφής δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Τι υπάρχει λοιπόν πίσω από αυτό το γεγονός. Στην έκθεση μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά στοιχεία από αυτού. Θέλω όμως να επισημάνω μόνο λίγα θέματα και πολύ γρήγορα. Προφανώς αυτά που είπα σχετικά με την θέση των ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει άμεσες επιπτώσεις και στο μισθολογικό στοιχείο σχετικά με τα δύο φύλλα. Βεβαίως δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένας αυτόματος ε, μηχανισμός ε, και αυτόματος, αυτόματες επιπτώσεις ε, στα δύο φύλλα. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι πιο σημαντικό. Αυτό που πολλοί το αποκαλούν διακριτική μεταχείριση. Στην έκθεση που αφορά στην μισθολογική εξέλιξη και στην κατάσταση των γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο υπάρχει μια πολύ περίπλοκη σχέση. Μπορείτε να ανατρέξετε στην ομιλία μου να τα δείτε, όμως θα ήθελα στην προφορική μου ομιλία να επισημάνω ένα θέμα το κόστος απόκτησης παιδιού. Αυτό έχει σχέσεις και επηρεάζει την αγορά εργασίας. Αυτό λοιπόν επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες. Για τις γυναίκες το να αποκτήσουν παιδί συνεπάγεται κόστος. Και αυτό το κόστος μετακυλείεται στις μισθολογικές τους αποδοχές υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο να αποκτήσουν οι γυναίκες παιδί και στις διακριτικές μεταχειρήσεις που υφίστανται σε μεστολογικό επίπεδο. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής. Το τελευταίο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε με τους συνεργάτες μου είναι το κατά πόσο να είναι κανείς ε, συνδικαλισμένος μπορεί να επηρεάσει και αυτό τους, τις ε, αποδοχές. Ξέρουμε ότι όσον αφορά ε, τις οικιακές βοηθούς αυτές δεν είναι συνδικαλισμένες και κατά κανόνα εργάζονται με μαύρη λατρέα μορφή εργασίας. Πάντως ε, θέλω να σας πω ότι τα στοιχεία που υπάρχουν ε, δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα. Αυτά που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, δείχνουν ότι το να εργάζεται κανείς σε ένα τομέα όπου υπάρχει έντονος συνδικαλισμός, αυτό ε, τελικά οδηγεί σε προστασία των αποδοχών. Υπάρχουν σαφώς διαφορές, μπορεί κανείς να προβεί στις ε, σχετικές αναλύσεις ε, και να διαπιστώσει ότι αυτό ισχύει κυρίως για τον δημόσιο τομέα και λιγότερο για τον ιδιωτικό. Και τώρα φτάνω στην τελευταία διαφορά την οποία έχω ελέγξει εγώ και πιστεύω ότι είναι μια διαφορά την οποία πρέπει να συγκρατήσουμε. Σας την ε, επισημαίνω ιδιαίτερα αυτή τη διαφορά. Είναι μια διαφορά που εμφανίζεται λιγότερο αλλά έχει μεγαλύτερη βαρύτητα έχει σχέση με την ηλικία αλλά έχει σχέση και με διάφορες δυναμικές που αναπτύσσονται στην αγορά εργασίας. Αναφέρομαι στις συντάξεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει σώρευση εργάσιμων ετών και από εκεί εξαρτάται η ε, σύνταξη την οποία παίρνουμε στα διάφορα κράτη-μέλη. Παραμένει όμως το γεγονός ότι αν τελικά κάνουμε τις, ε, τους υπολογισμούς με βάση τους μισθούς ε, που ε, χωρίζονται αυτή τη στιγμή, η διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες είναι περισσότερο από διπλάσια σε σχέση με τις αποδοχές της ενεργού ζωής. Υπάρχει λοιπόν αυτό το στοιχείο στις συντάξεις και εδώ διαπιστώνουμε μία σαφή επιδείνωση ε, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες σε πιο προχωρημένη ηλικία. Είναι σαφές, ε, μάλλον εντάξει ισχύει το ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο, έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, αλλά αν θέλετε ο μόνος τρόπος ε, για να προστατευτούν οι γυναίκες είναι ακριβώς να βρεθούν κάποιες δίκαιες ρυθμίσεις. Αναφέρομαι κυρίως στις γυναίκες που έχουν χάσει τον άντρα τους. Όλα αυτά, όπως σας είπα, έχουν και πάλι άμεση σχέση με την απόκτηση παιδιού. Οι γυναίκες έχουν λιγότερα αιτία εργασίας, ακριβώς λόγω αυτού του γεγονότος. Και έχει <clears throat> διεξαχθεί μια θαυμάσια μελέτη από το Network Canada, από τους συναδέλφου μου, είναι μια ε, μελέτη την οποία έχουν εκπονήσει άλφη από την Γενική Διεύθυνση ε, για θέματα δικαιοσύνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι από εκεί εξάγεται το συμπάρασμα ότι υπάρχει πλήρης και άμεση διασύνδεση ανάμεσα στις σταδιοδρομίες ε, που, των γυναικών που παρουσιάζουν ε, κάποιες διακοπές, ανάμεσα σε αυτό και στις ε, τελικές τους συνταξιωτικές απολαβές. Εγώ λοιπόν έχω φτιάξει έναν πίνακα από την έκθεση και τη μελέτη ε, στην, την οποία σας ανέφερα και εκεί βλέπετε ότι στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν βέβαια διαφορές όσον αφορά αυτές τις διακοπές που εμφανίζονται στις ε, σταδιοδρομίες των γυναικών. Ε, και θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου αναφερόμενη κυρίως σε, σε κάποιες προκλήσεις έχοντας κατά νου αυτές τις αλλαγές, τις νέες διαδρομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα ήθελα να έχουμε κατά νου ένα ρόδινο μέλλον και εδώ εμπνεύστηκα από ένα από το New Deal του Ρούσβελτ μετά την μεγάλη κρίση στην Αμερική. Τώρα ίσως ε, και εμείς να βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση που βιώσαμε ποτέ ως χώρες της δύση Είναι λοιπόν μια θαυμάσια ευκαιρία την κρίση αυτή να την εκλάβουμε ως μια νέα αρχή για την ισότητα των δύο φύλων. Σας ανέφερα τα αίτια και σας είπα γιατί πρέπει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είναι γνωστό ότι επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα ισότητας των δύο φύλων, αναφέρει ότι αν τελικά επενδύσουμε σε ε, θέματα που λαμβάνουν υπόψη τους ε, την ισότητα των δύο φύλων, όλα αυτά δηλαδή που εντάξει παρουσίασα, τότε η Ευρώπη θα μπορούσε να παρουσιάζει ανάπτυξη μεγαλύτερη ανάπτυξη κατά 2,4% από αυτήν που θα παρουσιάσει έτσι και αλλιώς μέχρι το 2030 θα υπάρξει αναμφίβολα μία βελτίωση από την ανάπτυξη που μπορεί κανείς να επιτύχει μέσα από διαφόρων ειδών ε, επενδύσεις και αναφέρομαι στο πακέτο ε, των κοινωνικών επενδύσεων ε, το οποίο παρουσιάστηκε κατά διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας και ακόμα περιμένουμε να δούμε μια ικανοποιητική ανάλυση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το πακέτο αυτό. Πρέπει λοιπόν να βαδίσουμε προς ένα νέο ροζ ε, deal, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, γιατί κατά την άποψή μου αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί, τουλάχιστον για τη δική μου τη χώρα. Τι πρέπει να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα, να υπάρξουν επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές που θα προκαλέσουν την απασχόληση, που θα ενθαρρύνουν ε, την ε, πρόσληψη γυναικών με δεξιότητες. Εγώ αναφέρουμε πάντα σε αυτά τα θέματα, να ληφθούν μέτρα που να έχουν σχέση με τη μέρημνα για τα παιδιά. Ε, δαπάνες για παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς, ε, για δημοτικά σχολεία, να ε, γίνουν επενδύσεις και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει ο στόχος της Βαρκελόνης. Φαντάζομαι θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Εκεί υπολείπονται ακόμα πολλές επενδύσεις, όχι όμως μόνο για να εγγυηθούν εγγυηθούμε την απασχόληση των ήδη των γυναικών που εργάζονται, αλλά και να εισέλθουν και νέες στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες έχουν πάρα πολλές δεξιότητες, μιλάμε για πολλές γυναίκες πτυχιούχους, άρα δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καλή ποιοτική μορφή απασχόλησης και όχι με την εκμετάλλευση. Θεωρώ λοιπόν ότι προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ε, εργασίας για τις γυναίκες που βρίσκονται σε, ήδη σε απασχόληση και για εκείνες που θα ε, βρουν θέση εργασίας. Αναφέρομαι εδώ σε νέες γυναίκες. Αναφέρομαι κυρίως στους ε, σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να παίξουν ρόλο και θα ήθελα να κλείσω σιγά σιγά Αναφέρομαι στις ε, εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια τα οποία εκπροσωπείτε και με τα οποία συνεργάζεστε. Όλοι αυτοί ε, θα πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσεις και τα λέω αυτά στην έκθεσή μου να αναλάβουν δεσμεύσεις για την εφαρμογή σωστών φορολογικών πολιτικών που θα ευνοούν την απασχόληση γυναικών. Ε, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ε, τα ε, φορολογικά μέτρα θα πρέπει να αφορούν γενικά την οικογένεια αλλά και τις γυναίκες πιο συγκεκριμένα. Οι γυναίκες ε, πολλές φορές δυστυχώς ε, εξαρτώνται από τους breadwinners, από αυτούς ε, που φέρνουν τα χρήματα στο σπίτι, που κατά κανόνα στις ε, χώρες μας είναι οι άντρες. Κατόπιν θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα επιδόματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις γυναίκες, βεβαίως και έχοντας κατά νου τις ε, ε, συνθήκες απασχόλησης και τις ε, συμβάσεις που σας ανέφερα στην αρχή που αφορούν ειδικά τις γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει κάνει πολλές φορές, αλλά σας καλώ να το ξανακάνετε. Να δρομολογήσει, να αναζητήσει αυτό το New Pink Deal με στόχο να αρτούν οποιασδήποτε στρεβλώσεις υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Αυτό βεβαίως πρέπει να γίνει με νόμιμο τρόπο. που και σε αυτόν τον τομέα υπολείπονται, κατά πολλά, υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά που αφορούν στις γυναίκες και κυρίως στις νέες γυναίκες οφείλουμε να αναζητήσουμε τη διαφάνεια και οφείλουμε πάνω απ' όλα να ενισχύσουμε αλλά και να υπεραμεινθούμε των θεσμών ίσων ευκαιριών που λόγω της κρίσης κινδυνεύουν οι θεσμοί αυτοί. Ε, υπάρχει μια τάση να αντιμετωπίζονται ως πολυτέλεια. Και κλείνω ε, προσπαθώντας ε, να συνδεθώ και με την προηγούμενη ομιλήτρια. Και θέλω να πω το εξής. Σαφώς και είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση που αναδείχθηκε προηγουμένως από την προηγούμενη μιλήτρια. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι, όπως σας είπα, να ε, προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τους δείκτες που δείχνουν τις διαφορές και το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Αυτοί οι δείκτες πρέπει να ενταχθούν σε διάφορες πολιτικές. Εγώ στη δική μου την έκθεση αναφέρω ότι γίνεται πράγματι μια πάρα πολύ καλή δουλειά ε, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή να λάβει υπόψη της ε, αυτά τους δείκτες και αυτές τις μελέτες που υπάρχουν. Υπάρχει ο δείκτης ε, περί ίσων ευκαιριών ε, που έχει εκπονηθεί και αυτό είναι νομίζω σημαντικός δείκτης που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ε, ευχαριστούμε πολύ αξιότιμη κυρία καθηγήτρια. Είναι ένα θέμα που μας συναρπάζει όλους και όλες. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεισφορά σας. Έχει έρθει λοιπόν η στιγμή να πάρουν το λόγο τα μέλη της Επιτροπής μας. Εάν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ να τις υποβάλλετε. Υπάρχουν ερωτήσεις για την κυρία Κόρση, καταρχάς η κυρία Χέντ και στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Σας παρακαλώ να είστε σύντομες και σύντομοι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Η κυρία Χέντ, εσείς πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι νιώθουν απογοητευμένοι. Πόσο μάλλον που πέρασε και το καλοκαίρι. Ωστόσο, στην προεκλογική εκστρατεία στη Σουηδία πάρα πολλές μέρες αφιερώθηκαν ε, ε, στο θέμα αυτό. Ήταν ένα θέμα πολύ ψηλά στην ε, πολιτική ημερήσια διάταξη. Είναι πολύ δυστυχές το γεγονός ότι έχει φτάσει και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος του 2014 και ακόμα τέτοια πράγματα συζητάμε και κάθε χρόνο πρέπει να προτείνουμε λύσεις σε θέματα τόσο σημαντικά, τόσο μεγάλα, τόσο περίπλοκα, όπως είναι π.χ. οι συντάξεις. Όλο αυτό έχει να κάνει με τις ίσες ευκαιρίες σε όλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής. Στη Σουηδία οι γυναίκες ε, καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου κερδίζουν 6 εκατομμύρια λιγότερο από ότι οι άνδρες σε αντίστοιχη απασχόληση. Είναι τεράστιο το μισθολογικό χάσμα. Πρέπει να βοηθούμε τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, κοινωνική πολιτική χωρίς να κλείσουμε αυτό το χάσμα, χωρίς να το γεφυρώσουμε. Πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα τώρα. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν ήδη από τώρα. Μιλούμε για όλα αυτά εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει έρθει πλέον η ώρα να περάσουμε στην πράξη. Η οδηγία για παράδειγμα για την άδεια μητρότητας είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος οι περισσότερες γυναίκες να αποκτήσουν περισσότερη απασχόληση πρέπει να έχουν όλες τις ίδιες ευκαιρίες απασχόλησης όπως και οι άνδρες, όπως και τον ανδρών. Και έτσι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το κράτος πρόνοιας κατά 11% και σε άλλες χώρες κατά 14% και 15%. Τα νούμερα αυτά είναι εξαιρετικά απογοητευτικά και μάλιστα εν έτη 2014. Ευχαριστώ ο κύριος Μαρίνο Πίντο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να, να συμφωνήσω με την ε, ομιλήτρια αλλά να κάνω και μερικά σχόλια και προτάσεις για τους λόγους χειροτέρευσης της κατάστασης των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχει μια σημειώνεται κρίση και σε τέτοιες περιπτώσεις τα πρώτα θύματα είναι οι γυναίκες. Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μου και αλλού. Γενικά οι γυναίκες ασχολούνται οικιακά, απασχολούνται οικιακά και πληρώνονται πολύ λίγο και συχνά πρέπει να διαλέξουν αν θα έχουν οικογενειακή ζωή και παιδιά ή επαγγελματική καριέρα από τη στιγμή που έχουν παιδιά δεν μπορούν πια να απασχοληθούν. Είναι κάτι πολύ σοκαριστικό. Στην Πορτογαλία το Opus δεν κυριαρχεί στην κοινωνική ζωή και εκκλησιαστικές οργανώσεις γενικότερα δεν απασχολούσαν γυναίκες λόγω του κινδύνου εγκυμοσύνης και μητρότητας. Αυτά έχουν αλλάξει χάρη στις επικρίσεις της κοινή γνώμης. Η Κομισιόν λοιπόν ετοιμάζεται να ετοιμάσει την καινούρια επιτροπή όπου θα υπάρχουν πολύ λίγες γυναίκες και αυτό είναι σοκαριστικό και θα ήθελα να κάνω εδώ μία έκκληση να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταψηφίσουμε αυτή την Κομισιόν ακόμη και αν αυτό δεν συμφωνεί με την πολιτική μου ομάδα. Εγώ προέρχομαι από χώρα όπου ο πληθυσμός είναι κυρίως καθολικός. Ας ζητήσουμε λοιπόν από την Καθολική Εκκλησία και άλλες εκκλησίες να μιλήσουν για αυτό το πρόβλημα. Στη χώρα μου υπάρχει πολύ μεγάλη λατρεία της Παναγίας της Φατίμα Έχω λοιπόν αναρωτηθεί πολλές φορές και ζήτησα, ρώτησα επισκόπους, είναι λογικό να έχουμε αυτή τη λατρεία της Παναγίας της Φατίμα, μιας γυναίκας δηλαδή, ενώ η πολιτική που εφαρμόζουμε εμποδίζει τις γυναίκες ακόμη και να μεταλάβουν των αχράντων μυστηρίων επειδή είναι γυναίκες. Στους καθολικούς γάμους το κείμενο που πρέπει να διαβάσει μια γυναίκα κατά την τελετή του γάμου είναι διαφορετικό από το άντρα. Οι γυναίκες πρέπει να δίνουν όρκο υπακοής, όχι πίστεως, υπακοής. Άρα είναι κτήμα του άντρα η γυναίκα. Αυτό είναι πολιτισμός που προέρχεται απευθείας από το ρωμαϊκό δίκαιο, από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και ισχύει ακόμα για την οτροπία, στην οτροπία πολλών. Σας προτείνω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και τα κράτη-μέλη της χωριστά να υποστηρίξουν όλες τις επιχειρήσεις και ιδιωτικές που, που λέγω θα σέβονται ορισμένες ποσοστώσεις της προσλήψης γυναικών. Οι 50-50 δηλαδή της 100. Εξάλλου κάποιος επαναστάτης έλεγε ότι οι γυναίκες φέρουν το ίμιση του βάρους τους κατά την εγκυμοσύνη και δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς ή τη δυνατότητα μάλλον εμείς οι άντρες να κάνουμε κάτι τέτοιο. Πόσοι άντρες θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την ανατροφή ενός παιδιού. Στην Ένωση πρέπει να καταπολεμήσουμε, να καταπολεμήσουμε λέγω να καταπολεμήσουμε την τάση, την, τον πειρασμό να εφαρμοστούν μέτρα και πολιτική που να μην προωθούν την ισότητα των φύλων. Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ ε, πολύ ε, την εισηγήτριά μας για όλα αυτά που μας είπε. Προηγουμένως μας είπατε ε, τι δυσκολίες παρουσιάζει η αγορά εργασία κυρίως ε, για τις γυναίκες. Επιτρέψτε να σας κάνω μία ερώτηση κάτω από διαφορετικό πρίσμα. Κοιτάξτε, η αγορά εργασίας και ο κόσμος εργασίας τα τελευταία χρόνια άλλαξε ριζικά λόγω της ψηφιοποίησης. Σήμερα λοιπόν ε, διαπιστώνουμε ότι μπορεί κανείς ε, να εργάζεται σε τελείως διαφορετικό χώρο από εκεί που είναι το αντικείμενο της εργασίας. Ας πούμε εγώ γνωρίζω πολλές γυναίκες που λόγω της ψηφιοποίησης δουλεύουν σε ένα κάποιο χώρο εργασίας, κάποιες ε, τελείως διαφορετικές ώρες από ό,τι πιστεύει κανείς. Άρα δηλαδή θεωρώ ότι αυτό ε, έχει και προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες ε, για τις γυναίκες για να εργαστούν, να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα και θέλω να σας ερωτήσω, αυτό το ερευνήσατε Ποιες είναι οι ευκαιρίες που έχουν προκύψει στο χώρο της εργασίας για τις γυναίκες λόγω της ε, ψηφιοποίησης. Και εντάξει, ξέρω ότι αυτό δεν θα σας το είχαμε πει να το ελέγξετε στο πλαίσιο της μελέτης, αλλά κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο να ασχοληθούμε με αυτό που σας λέω, δηλαδή να μην κοιτάμε μόνο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, να κοιτάμε και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για αυτές, να δούμε πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε να ε, αδράξουν αυτές τις ευκαιρίες να μην τα περιμένουν όλα από το κράτος. Γι' αυτό λοιπόν κυρία ε, καθηγήτρια θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσον ελέγξατε αυτές ε, τις ευκαιρίες ε, που προσφέρονται για μας τις γυναίκες λόγω της παγκοσμιοποίησης και λόγω της ψηφιοποίησης. Ευχαριστώ. κυρία Αρένα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκτύπησα ιδιαιτέρως ε, την παρέμβαση της ε, κυρίας καθηγήτριας, η οποία ήταν εξαιρετικά αποφασιστική θα έλεγα. Τρία είναι τα σχόλια που θα ήθελα να κάνω. Πρώτον, ο ρόλος των συνδικάτων. Είπατε ότι είναι μικρότερο το μισθολογικό χάσμα στο δημόσιο τομέα, γιατί η συνδικαλιστική εκπροσώπηση είναι πιο παρούσα, πιο ισχυρή. Ίσως, είναι η απάντησή μου. Ωστόσο, στο δημόσιο τομέα κωδικοποιούνται καλύτερα τα καθήκοντα, τα αξιώματα ή θέσεις και άρα σε μια πολύ πιο σαφή η ιεράρχηση, είναι πιο δύσκολο να υπάρχουν ζώνες διαπραγμάτευσης τις οποίες να αξιοποιούν περισσότερο οι άνδρες παρά οι γυναίκες. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο με τις ειδικαλιστικές οργανώσεις για να έχουμε περισσότερη κωδικοποίηση των θέσεων εργασίας έτσι ώστε να μειωθούν οι γκρίζες ζώνες τις οποίες γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο οι γυναίκες από ότι οι άνδρες και αυτό το γνωρίζουμε έχει φανεί ιστορικά. Σήμερα λοιπόν με την κρίση το, θέμα που, το ερώτημα που τίστε είναι το εξής. Γίνεται αναδιάρθρωση και στα συνδικάτα, ε, αναδιάρθρωση και στην ε, εκπροσώπηση των αρένων και άρα ε, γενικά έχει μειωθεί το ενδιαφέρον για την προώθηση των σκοπών των, της ισότητας των φύλων. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδουλέψουμε έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε εκ νέου τα συνδικάτα για να υπάρξει πραγματική ισότητα γυναικών και ανδρών στο χώρο εργασίας, κάτι που θα επιτευχθεί με καλύτερη κωδικοποίηση και περιγραφή των θέσεων των αξιωμάτων των λειτουργιών. Μπορεί να μην συμφωνούν όλοι και το γνωρίζω. Στη χώρα μου όμως η πολιτική διαβούλευση, ε, η κοινωνική διαβούλευση είναι κάτι το πολύ σημαντικό και τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο θετικά όταν είναι προϊόν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έρχομαι τώρα στο τρίτο θέμα που είναι η γυναίκα επιχειρηματίας, η δυνατότητα για τις γυναίκες να δημιουργήσουν τη δική τους απασχόληση. Πολύ συχνά όταν μιλούμε για γυναίκες επιχειρηματίες εννοούμε γυναίκες φτωχές περιοχές επιχειρηματίες και δηλαδή θέλουμε να φύγουν από την ε, συλλογική προστασία, από μια συλλογική πλαισίωση γιατί είναι γυναίκες και φτωχές και θέλουμε να ασχοληθούν επιχειρηματικά με κάτι ε, έτσι ώστε να μείνουν μόνες τους πλέον και να το παλεύουν. Υπερασπίζομαι βέβαια τη δημιουργία και τη δημιουργικότητα των γυναικών. Εάν όμως ε, από το παράθυρο και δια της πλαγίας οδού θέλουμε τις γυναίκες τις φτωχές να τη βγάλουμε από το κοινωνικό πλαίσιο υποστήριξης για να αποκτήσουν υποτίθεται κάτι δικό τους και να το δουλέψουν, ε, είμαι κατά γιατί ε, αυτό θα τις αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο. Τέλος, Μιλήσατε για τις κοινωνικές πολιτικές, για τις συλλογικές υποδομές, π.χ. φύλαξη παιδιών κτλ. Τα στατιστικά στοιχεία μας μαθαίνουν ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τη δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή επιλέγουν π.χ. μερική απασχόληση γιατί έχουν μια μισθολογική ε, ανταμοιβή και το κάνουν γιατί κυρίως οι μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί είναι οικογένειες που ο είναι γυναίκα και το καθεξής. Με το σύμφωνο Σταθερότητας ως χώρα τελικά πήραμε μέτρα για τη μείωση των κοινωνικών δαπανών. Στις μελέτες σας έχετε μελετήσει εάν υπάρχει αντίκτυπος του Συμφώνου Σταθερότητας και αν έχει αυξήσει τη φτώχεια των γυναικών και τις έχει εμποδίσει από το να προσχωρήσουν στην αγορά απασχόλησης. Και επόμενο θέμα, οι συντάξει. Πολλοί λεπτό το ζήτημα πράγματι. Ωστόσο, στην Ευρώπη, σε πολλά κρατημέλη, υπάρχει η τάση να ενθαρρύνουμε την πρόσβαση στο δεύτερο ή τον τρίτο πυλώνα, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο. Δηλαδή, ο δεύτερος ε, το, ε, πυλώνας ενθαρρύνει τους πιο πλούσιους κλάδους και ο τρίτος πυλώνας ενθαρρύνει τους πιο ψηλούς μισθούς. Άρα όχι τις γυναίκες σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Άρα ε, έτσι όπως έχει στραφεί το συνταξιδοτικό σύστημα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και οι κατευθύνσεις που παίρνει δεν είναι κάτι που θα κάνει τη θέση της γυναίκας ακόμα πιο ευπαθή και αβέβαια. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Η κυρία Βάρντ, η Ευχαριστώ πολύ και εγώ είχα ζητήσει το λόγο, αλλά μάλλον δεν με είδατε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Καταρχήν και εγώ να σας ευχαριστώ θερμά για το ότι τα ξεκαθαρίσατε λιγάκι αυτά που λέγονται, ότι οι άντρες κυρίως πλήττονται από την κρίση. Δεν ισχύει αυτό. Αλλά όπου και αν βρισκόμαστε, πράγματι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παρουσιάζουν αυτά τα στατιστικά δεδομένα. Εγώ θεωρώ όμως ότι αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα κοινική. Κοινική προσέγγιση που εγκυμονεί τον κίνδυνο ε, τα αιτήματα των γυναικών να περιφερειοποιούνται και κυρίως να εξανδραποδίζονται από τις οικονομικές συζητήσεις. Αυτό όμως και πάλι δείχνει το πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύσει με διαφορετικούς τρόπους και να αλλοιώσει στατιστικά δεδομένα. Επιτρέψτε μου και άλλη μια ερώτηση, στατιστικής φύσεως. Αναφερθήκατε στο θέμα της ε, μερικής απασχόλησης. Εγώ προέρχομαι από την Αυστρία. Σε εμά το θέμα αυτό είναι φλέγον, διότι η αύξηση της απασχόλησης, του ποσοστού απασχόλησης ε, στις γυναίκες οφείλεται καθαρά και μόνο στη μερική απασχόληση. Κάτι που εμείς το βλέπουμε με πολύ επικριτικό πνεύμα. Και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, εσείς έχετε κάποια στατιστικά δεδομένα ε, που να δείχνουν τις επιπτώσεις σε άνδρες και γυναίκες σε κατάσταση όμως πλήρους απασχόλησης. Ε, έχετε κάποιες, ε, κάποια μισθολογικά στοιχεία ή έχετε έτσι γενικότερους φύσεως διαπιστώσεις ότι οι γυναίκες υφίστανται περισσότερες αρνητικές συνέπειες από τους άνδρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια ως προς την έρευνα, τη διάσταση της έρευνας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύονται οι διακρίσεις. Καλό θα είναι λοιπόν να μην μιλούμε μόνο για τη διαφορετική κατάσταση ανδρών και γυναικών, αλλά θα πρέπει να δούμε και την κατάσταση των γυναικών στις ε, υποτιθέμενες χώρες μέλη πρώτης κατηγορίας και την κατάσταση των γυναικών στις υποτιθέμενες χώρες μέλη δεύτερης κατηγορίας, γιατί αυτό υπάρχει ήδη. Ε, π.χ. Ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις, ε, με αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, ας ε, θέσουμε αυτό το παράδειγμα με μια, μιας αυστριακής ε, υπαλλήλου που συγκρίνεται με μια Ουγγαρέζα υπάλληλο ε, σε αυτό το την πολυεθνική με αλυσίδα καταστημάτων λιανικής και το καθεξής. Όλα θα πρέπει να γίνουν έρευνες δηλαδή και σε αυτά τα πεδία και μελέτες. Από εκεί και πέρα Πράγματι τα συνδικάτα είναι ισχυρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από ορισμένους κλάδους. Λέτε, μπορεί αυτό να ισχύει στις δυτικές χώρες μέλη, αλλά σε καμία περίπτωση ε, δεν ισχύει σε άλλες χώρες μέλη που θεωρούνται υποδέστερες δεύτερης κατηγορίας και τις οποίες ε, ουσιαστικά υπάρχει αντιμετώπιση ως αν επρόκειτο για απικίες. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, μπορεί να έχει υπάρξει και απαγόρευση να συζητά κανείς για αυτά τα θέματα. Να δούμε και το θέμα των γυναικών μικροεπιχειρηματιών. Γυναίκες που έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή εισραίουν τα ξένα αγαθά πάλι έρχονται στο προσκήνιο οι πολυεθνικές. Είναι αδύνατο να ανταγωνιστεί κανείς τις εταιρείε κολοσσούς. Όλα αυτά είναι καθόδη ζητήματα, δύσκολα ζητήματα, πρέπει να γίνει έρευνα πάνω σε αυτά και πρέπει να δούμε και ε, το ότι όταν θέλει κάποιος να φτιάξει μια οικογένεια, το βάρος ε, ε, δυσανάλογα το, το επομίζεται η γυναίκα το γεγονός ότι, για παράδειγμα, οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ε, σε πολλούς απαραίτητους φορείς ή το, ότι, το γεγονός ότι υπομίζονται μονο στο βάρος της ανατροφής του παιδιού όταν ή αν επέλθει το διαζυγείο είναι ε, θέματα που αυξάνουν την πιθανότητα το συγκεκριμένο παιδί ή το εκάστοτε παιδί να ε, βιώσει σε καθεστώς φτώχειας. Για κάθε, για κάθε παιδί που ζει σε καθεστώς φτώχειας υπάρχει και μια γυναίκα πίσω του που ε, ζει και εκείνη σε καθεστώς φτώχειας και πρέπει να θυσιάσει πάρα πολλά. Οι πάρα πολλές από αυτές ε, δεν τρώνε και πεινούν προκειμένου το λιγοστό φαγητό να το δώσουν στο παιδί τους. Και πρέπει να δούμε και πώς συμπεριφέρεται το, το κράτος υπ' αυτή την έννοια. Όλα αυτά έχουν σχέση με την οικονομική ανεξαρτησία. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Έχει ολοκληρωθεί ο γύρος ερωτήσεων. Η τελευταία κυρία Βάρτ, παρακαλώ. Um, σας ε, ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο ομιλίες. Εγώ λοιπόν αισθάνομαι ότι υπάρχει επίθεση από πολλά μέρη και είναι δύσκολο να δει κανείς ε, περί τίνος ακριβώς πρόκειται σχετικά με τα συνδικάτα. Γνωρίζουμε ότι τα συνδικάτα δέχονται επιθέσεις. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν ε, να εγγυηθούμε ότι αυτή θα είναι η θέση που θα προβληθεί γιατί υπάρχει σαφώς το θέμα της ε, λιτότητας. Είδα στα στατιστικά δεδομένα που προβάλλατε ότι το χειρότερο χάσμα είναι σε θέματα εξουσίας. Σωστά το λέω. νομίζω υπάρχει ένα χάσμα περίπου της τάξης του 30%. Αν λοιπόν αυτό ισχύει, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα συσχετισμό ανάμεσα στην έλλειψη αρμοδιοτήτων και εξουσίας που έχουμε ε, και που οδηγεί στο ότι ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά σε σχέση με, για τη θέση των γυναικών απέναντι στην Επιτροπή. Αυτό να το συσχετίσουμε με την εκπροσώπηση, αυτά που θα πει η δική μας η Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά τα οποία είπατε σήμερα ε, νομίζω εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο που συζητάμε. Ήθελα απλά να διπλοτσεκάρω, γιατί είδα στα στατιστικά δεδομένα ε, τι το θέμα των αρμοδιοτήτων. Και αυτό μας δίνει εμάς τη δυνατότητα να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε περαιτέρω τις απαραίτητες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βάρντ Η Ward. Όπως είπε και η κυρία και όπως ακούσαμε και από τις ε, παριστάμενες, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η παρουσίαση για την άδεια μητρότητα, την οδηγία για την άδεια μητρότητα, η οποία είναι και εξαιρετικά σημαντική, μπορεί να γίνει το απόγευμα. Και άρα θα ολοκληρώσουμε έχοντας ακούσει τις καθηγήτριες οι οποίες θα απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Και αν έχουμε χρόνο και μείνει ε, λίγος χρόνος, τότε θα ασχοληθούμε με την ε, οδηγία για την ε, άδεια μητρότητα. Ιδαλλιώς θα ασχοληθούμε μαζί της το απόγευμα. Σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας τέθηκαν, κυρία Κόρση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που μου δίνει τη δυνατότητα να απαντήσω γιατί πάντα είναι μεγάλη χαρά το να μπορεί κανείς ε, να ε, έρχεται σε συζήτηση με πολιτικούς παράγοντες. Λοιπόν, τα σημείωσα αυτά που μου είπατε. Τώρα, αν κάτι μου ξέφυγε, ζητώ συγγνώμη. Σημείωσα όμως αυτά που μου φάνηκαν τα πιο κρίσιμα, τα πιο επίγοντα. Λυπάμαι που έφυγε η Ευρωβουλευτής από τη Σουηδία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα και εγώ να πω ότι υπάρχει τεράστια ένταση και απογοήτευση και από δική μας πλευράς. Ήρθα και εγώ εδώ στο Κοινοβούλιο για να καταγγείλω το ότι δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος. Όμως το όνειρο που θέλησα ε, σε εισαγωγικά να σας πουλήσω δεν είναι ένα τυχαίο όνειρο, είναι κάτι πάνω στο οποίο δουλεύουμε και αφορά την νέα εξέλιξη που πρέπει να λάβει η ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι πλέον μια ευκαιρία που δεν πρέπει να την χάσουμε καθώς θα τελειώνει η κρίση είναι μια ευκαιρία που αφορά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε οικονομικό επίπεδο, αλλά ε, υπάρχουν και άλλα θέματα που και άλλα μέτρα πρέπει να ληφθούν, ε, γιατί βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Γι' αυτό και αναφέρθηκα στο New Deal του Ρούσβελτ που άφησε ανεξίτηλα ε, ίχνη στην αμερικανική πολιτική. Αυτό λοιπόν ε, είναι το όνειρο. Για να υλοποιήσει κανείς ένα όνειρο, προφανώς και πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται. Αυτό νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό ότι πρέπει να σκεφτεί πίεση κυρίως ε, για θέματα που αφορούν ε, στη γονεϊκή άδεια. Ε, λυπάμαι που έφυγε η συνάδελφος, αλλά ίσως μας ξαναδοθεί ευκαιρία για να συζητήσουμε. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά που σημείωσα, κυρίως σε αυτά που είπε ο συνάδελφος από την Πορτογαλία, Θέλω να πω το εξής, ότι εγώ ε, ανησυχώ για το ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται χωρίς δίκες απολαβές. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Πορτογαλία, αφορά και πολλές άλλες ε, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Βλέπουμε ότι ε, ακριβώς λόγω αυτού του γεγονότος ε, προκύπτει και το θέμα της ε, μετανάστευσης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Ευρώπη. Υπάρχει εργασία των γυναικών που δεν αμείβεται και με πολύ μεγάλη χαρά θα ακούσω σήμερα το απόγευμα την έκθεση και την ομιλία που θα γίνει επ' αυτού του θέματος. Αυτά που θα ακούσετε σήμερα, όλες αυτές οι συγγύσεις διασυνδέονται μεταξύ τους και γι' αυτό το λόγο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας ε, να πούμε κάτι ξεχωριστό Δηλαδή ε, θα έπρεπε ίσως ε, να αναζητήσουμε κάτι καινούριο, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν τελείως διαφορετικά ε, επιχειρήματα από τους προηγούμενους ομιλητές. Τώρα, την Millennium Bank είναι μια τράπεζα στην Πορτογαλία, η οποία ασχολείται με την καταναλωτική πίστη και αυτό είναι κάτι το οποίο το σημείωσα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι για να επανέλθω λιγάκι στα στατιστικά δεδομένα, σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη η επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών είναι η μόνη περίπτωση που υπήρχε για τις νέες γυναίκες για να βρουν θέση απασχόλησης, κάποια απασχόληση, κυρίως πρώτη απασχόληση, που αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που αφορά κατά κύριο λόγο μόνο τους νέους. Υπάρχουν βέβαια κάποια ε, κάποιες περιπτώσεις στην Ισπανία που συζητήθηκαν πάρα πολύ από τη σχετική βιβλιογραφία. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε σχετικά με τις γυναίκες επιχειρηματίες ότι το θέμα είναι πολύ περίπλοκο. Πάω τώρα στο θέμα της τεχνολογίας. Αναμφίβολα σε ιδιαίτερα ε, τεχνολογικά εξελιγμένες επιχειρήσεις οι γυναίκες μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ε, τις ε, δεξιότητες τους. Αυτό δεν το είπαμε, αλλά να σας το πω τώρα ότι οι γυναίκες σε επίπεδο δεξιοτήτων ξεπέρασαν κατά πολύ τους άντρες κατά τα τελευταία έτη. Υπάρχουν ε, σχετικές ε, μελέτες που το ε, τεκμηριώνουν αυτό. Οι γυναίκες, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ καλές και έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες πλέον και κυρίως και στο θέμα της εκπαίδευσης. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν τόντι να εργαστούν σε διάφορους τομείς. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς εξακολουθούν να μην υπάρχουν πολλές γυναίκες σε ανώτατες τεχνολογικές θέσεις. Αυτό αφορά κυρίως ε, θέσεις ε, μηχανικών επιστημόνων, ειδικών επιστημόνων και θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ειδική έκθεση ε, η οποία έχει εξετάσει διάφορους ε, τομείς. Εκεί λοιπόν προκύπτει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ουσιαστική διακριτική μεταχείριση και οι γυναίκες δεν υπάρχουν σε πολλές θέσεις υψηλής τεχνολογίας. Υπάρχει κυρίως μια περίπτωση στη Φινλανδία. Θα θυμάστε ότι το 2008 το Υπουργείο Εργασίας στη Φινλανδία ε, διεξήγαγε μια, ε, μια εκστρατεία για να μην, υπάρχει, ε, μην υπάρχουν μισθολογικές διαφορές στη Φινλανδία. Αναφέρομαι στην περίπτωση της Νόκια. Και τότε ε, θα θυμάστε ότι αναφέρθηκε αυτή η περίπτωση για να ε, καταδειχθεί ότι υπάρχουν αυτές οι μισθολογικές διαφορές ε, στη Φινλανδία. Στη Φινλανδία, μια σκανδιναβική χώρα που προφανώς πολλοί από εμάς ζηλεύουμε και θα θέλαμε να ζήσουμε ακριβώς λόγω του ότι προσφέρει πάρα πολλέ ευκαιρίε η χώρα αυτή σε επίπεδο τεχνολογική εξέλιξη. Η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχει όμω κάτι άλλο που αφορά την ε, εξαποστάσεως εργασία. Προφανώς και είναι μια ευκαιρία αυτή σήμερα, αλλά μπορεί να είναι και παγίδα. Και εδώ ε, συνδέω αυτό που σας λέω και σε σχέση με την επόμενη ερώτηση που ετέθη, ε, διότι ε, το θέμα της ε, εργασίας εξ αποστάσεως ε, οδηγεί σε πολύ μεγάλη απομόνωση. Με αυτήν την μορφή απασχόλησης υπάρχει ο κίνδυνος κυρίως για τις γυναίκες που παράλληλα κάνουν και πάρα πολλές άλλες δουλειές που προσέχουν τους ηλικιωμένου, προσέχουν τα παιδιά τους. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κίνδυνος απομόνωσης που δεν είναι οικονομικό στοιχείο που όμως και αυτό επιβαρύνει πολύ την ε, ποιότητα της ζωής τους, πόσο μάλλον της εργασίας τους. Η επιχειρηματικότητα είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί σε βάθος. Ε, εγώ σας είπα ότι δεν έχω το χρόνο και και το χώρο για να εξετάσω όλο αυτό το θέμα, το δύσκολο θέμα. Η ε, γυναίκες ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενες. Και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία που και αυτή αξίζει τον κόπο να την εξετάσουμε. Εξακολουθεί να παραμένει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και επανέρχομαι στο θέμα της ζωής των γυναικών επιχειρηματιών. Ε, μια γυναίκα επιχειρηματία σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή πολύ συχνά εργάζεται 20 ώρες ε, το 24ωρο ε, γιατί παίρνει τη δουλειά στο σπίτι της, ε, ακόμα και το να είναι κανείς ε, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο, αυτό είναι σαν να είναι κανείς επιχειρηματίας, γιατί αν δεν έχει ουσιαστική πειθαρχία, καταλήγει στο να εργάζεται 20 ώρες το 24ωρο. Θέλω λοιπόν να σας πω γιατί μας είπατε ότι πρέπει να αναφέρουμε και τις βέλτιστες, βέλτιστες πρακτικές. Ε, στη Φιλανδία υπάρχει ένα παράδειγμα, ένα Ινστιτούτο, ένα συγκεκριμένος οργανισμός για τις γυναίκες ε, επιχειρηματίες. Ε, υπάρχουν λοιπόν στοιχεία που αναφορούν κυρίως και μόνο τις γυναίκες επιχειρηματίες. Είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα Μία γυναίκα λοιπόν, αν αισθάνεται άσχημα ή αν έχει προβλήματα στην οικογένειά της, ε, τότε ε, μπορεί να υπάρξει κάποιος άλλος που να την αντικαταστήσει. Αυτό είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερα αξιόλογο πείραμα που ε, έγινε. Σε μας θέλησαμε να ε, εφαρμόσουμε το ίδιο στο Βένετο ε, που είναι μια πολύ βιομηχανοποιημένη περιοχή στην Ιταλία. Δεν ξέρουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Δεν έχει γίνει η σχετική αξιολόγηση. Πάντως ε, ο ΣΕΒ ας πούμε της περιοχής Βέντο της Ιταλίας είναι διατεθειμένος ε, να εφαρμόσει τέτοιου είδους ε, πειράματα. Πάμε τώρα στο ρόλο των συνδικάτων που ετέθηκε αυτό. Σας είπα ότι αυτό δεν το έχω εξετάσει το θέμα σε βάθος. Απλά ανέτρεξα στη βιβλιογραφία που υπάρχει αλλά θέλω να, να ε, αναφερθώ σε μία παρεξήγηση. Δεν είναι αλήθεια ότι στο δημόσιο τομέα υπάρχουν μεγαλύτερες ισότητες γιατί εκεί είναι πιο έντονος ο συνδικαλισμός. Δεν ισχύει αυτό. Πάντως, πράγματι στο δημόσιο τομέα προστατεύονται εκ του νόμου τα συνδικάτα. Υπάρχει βέβαια κίνδυνος αποδυνάμωση των συνδικάτων. Και αυτό αφορά κυρίως ε, τους ε, τομείς που αντιμετωπίζουν ε, κρίση. Γιατί λόγω των νεοφιλελεύθερων αυτών τάσεων και εξελίξεων που επικρατούν, πολλοί τάσσονται υπέρ της κατάργησης των συνδικάτων. Ορισμένοι συνάδελφοι ε, που υποστηρίζουν τέτοιες ε, νεοφιλελεύθερες απόψεις τάσσονται υπέρ αυτού. Δηλαδή, αν τελικά η πλήρης ε, απελευθέρωση στην αγορά ε, μας οδηγήσει εκτός της κρίσης, προφανώς και αυτό θα σημαίνει ριζική αλλαγή του συνδικαλισμού. Αυτό βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη απειλή για το χώρο της εργασίας, κυρίως για την ισότητα των δύο φίλων. Γιατί τα συνδικάτα δεν μπορεί κανείς να γενικεύσει, ε, ποικίλει κατάσταση από χώρα σε χώρα, Υπάρχει το θέμα των μικρών επιχειρήσεων, που προφανώς εκεί δεν υπάρχει συνδικαλισμός. Μιλάμε, μιλάμε άρα για μεγάλες επιχειρήσεις όταν μιλάμε για συνδικαλισμό. Πάντως, είναι ένα θέμα που κατά την άποψή μου πρέπει να παραμείνει στη συζήτηση δεν ξέρω και δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ε, σχέσεις ε, και επαφές ε, με το συνδικαλιστικό κίνημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι λοιπόν σαφές ότι αναφέρομαι στην ε, Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων γιατί ε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να αξιολογήσω τα θέματα τα συνδικαλιστικά σε άλλες χώρες. Ε, Italia Welfare όπως αναφέρθηκε. Και εδώ ε, θέλω ε, να πω ότι υπάρχει δυστυχώς σε μία παρεξήγηση. Εγώ αναφέρθηκα στους ε, θεσμούς ε, παιδικής μέρημνας γιατί συνήθως μιλάει κανείς για τέτοιου είδους φορείς αλλά προφανώς εξίσου σημαντική είναι και η μέρημνα για την τρίτη ηλικία. Αυξάνεται μάλιστα το πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα. Πάρα πολλές γυναίκες ε, 30 έως 40 ετών ε, έχουν το καθήκον να ε, μεριμνούν όχι μόνο για τα παιδιά τους αλλά και για άτομα τρίτης ηλικίας διότι δυστυχώς ε, όπως σας είπα δεν υπάρχουν αρκετοί θεσμοί παιδικής μέριμνας. Και αυτό είναι ένα θέμα που επηρεάζει πάρα πολύ και τη Μέριμνα για την τρίτη ηλικία. Θέλω να επαναλάβω ότι οι γυναίκες πράγματι έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, ε, ζουν όμως χειρότερα. Άρα δηλαδή ε, και αυτές ε, κάποια στιγμή από άτομα τα οποία προσφέρουν μέρημνα εξελίσσονται σε άτομα που χρήζουν μέρημνας. Εδώ λοιπόν πρέπει να σημάνει συναγερμός και θα ήθελα να επαναλάβω το 2011 τότε έγινε λόγος για το Social Investment ε, Package ε, εκ μέρους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τότε γίνεται λόγος για τη δέσμη μέτρων, μέτρα τα οποία θα ήταν η άλλη πλευρά του νομίσματος της λιτότητας. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο θα έπρεπε να ληφθούν κάποια μέτρα για να εξισορροπήσουν τις αρνητικές συνέπειες. Ε, θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να απαντήσει τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι ακριβώς έγινε με αυτή την αξισορρόπηση των αρνητικών συνεπειών σε κοινωνικό επίπεδο. Υπάρχει, όπως σας είπα, αυτό το κοινωνικό πακέτο και ελπίζουμε ότι θα ανανεωθεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω. Τώρα, σας ευχαριστώ πολύ που αναφερθήκατε σε διάφορα στοιχεία. Προς ενημέρωσή σας θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια έκθεση ε, την, στο θέμα το συνταξιοδοτικό. Στις συντάξεις λοιπόν ε, πράγματι υπάρχουν ε, διάφορα στοιχεία που παρισφρίουν στο θέμα το συνταξιοδοτικό. Και θέλω να πω ότι υπάρχουν και προηγούμενες εκθέσεις και τώρα έρχομαι στο θέμα το οποίο έθιξε η συνάδελφος από την Ουγγαρία. Πράγματι υπάρχει το θέμα των μεταναστών. Εγώ δεν το έχω εξετάσει αυτό το θέμα των ε, μεταναστών ή μεταναστριών και των συντάξεων. Υπάρχει το θέμα της ε, δυνατότητας μεταφοράς συνταξιδιωτικών δικαιωμάτων. Αυτό το θέμα δεν το έχω θίξει. Και βλέπω ότι αυτό το θέμα το έθιξε η κυρία από την Ουγγαρία, αλλά άμα υπάρχουν και βουλευτές ε, από άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, προφανώς θα γνωρίζουν όλοι ότι ε, το θέμα αυτό αφορά όλες τις δικές σας τις χώρες. Βλέπουμε λοιπόν και ξέρουμε ότι υπάρχουν εργαζόμενες με πολύ χαμηλές απολαβές και είναι και πολύ δύσκολο να ε, ενταχθούν, να νομιμοποιηθούν οι εργαζόμενες αυτές. Όταν, εν πάση περιπτώσει, νομιμοποιούνται, κάποια στιγμή αρχίζουν να καταβάλουν τις εισφορές τους. Τα χρήματα αυτά των εισφορών των μεταναστών τελικά πού καταλήγουν. Κανείς δεν ξέρει πού ακριβώς καταλήγουν. Ακόμα και σε περιπτώσει ανθρώπων που έχουν θεμελιώσει συνταξιωτικό δικαίωμα, είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρει κανείς τα συνταξιωτικά του δικαιώματα. Πάρα πολύ δύσκολο για τις γυναίκες. Και σας λέω κυρίως στον χώρο των οικιακών βοητών, επειδή εκεί έχουμε κυρίως γυναίκες, στον τομέα αυτό εμφανίζεται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάντως, μιλάμε για άντρες, για γυναίκες, για ηλικιωμένα άτομα για μετανάστες και εάν ε, ήμασταν μία χώρα με περισσότερες εθνότητες θα έπρεπε οπωσδήποτε να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, και αυτό το στοιχείο. και ο ε, σεξουαλικός προσανατολισμός. Παρακαλώ μην το ξεχνάτε και αυτό, γιατί ορισμένα από αυτά που είπα για τους άντρες και τις γυναίκες, ορισμένα εξ αυτών δυστυχώς το βλέπουμε αυτό και στα στατιστικά δεδομένα, επιδεινώνονται και λόγω των σεξουαλικών προτιμήσεων και του σεξουαλικού ε, προσανατολισμού. Όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα, τα στατιστικά δεδομένα είναι σαφές. Δεν ξέρω, στην Ιταλία Υπήρχε ένα ποιητή. που λέει ότι η μισή από τους ε, Ιταλούς, ε, αν δει κανείς τα στατιστικά δεδομένα, δεν έχουν τίποτα να φάνε. Εξαρτάται δηλαδή πώς ακριβώς ε, ερμηνεύει τα στατιστικά δεδομένα. Στο θέμα των στατιστικών δεδομένων έχει υπάρξει πρόοδος. Υπάρχει ε, η φόρμουλα του Πεκίνου σχετικά με τους ε, δείκτες ε, και εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι στη δική μου τη μελέτη στη συνεργασία που είχα με το Ινστιτούτο Ίσων Ευκαιριών του Βίλνεους και στη συνεργασία μου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρομαι στο Συμβούλιο του Ιουλίου του 2014 όπου όπως σας είπα γίνεται αναφορά στο ότι θα πρέπει ε, στην Ευρώπη να επιληφθεί κανείς ε, περισσότερο με θέματα τα οποία ε, προέκυψαν στα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης του Πεκίνου. Ε, κοιτάξτε για το θέμα της ε, μερικής απασχόλησης. Αυτό δεν υπάρχει μόνο στην Αυστρία, υπάρχει και στη Γερμανία. Γενικά υπάρχει η ακούσια μερική απασχόληση η οποία δυστυχώς όμως προκύπτει όλο και περισσότερο λόγω της κρίσης. Εντάξει, υπάρχει κάποια απασχόληση αλλά όμως θα πρέπει κανείς να αξιολογήσει τις επιπτώσεις μακροπρόθεσμα. Ε, αυτοί που κερδίζουν 500-600 ευρώ ε, θα πρέπει κανείς να δει τι θα γίνει τελικά με αυτούς, με τα δικά τους τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Η μερική απασχόληση ε, δυστυχώς ε, αυτή τη στιγμή υποτιμάται. Προφανώς λοιπόν συμμερίζουμε τις δικές σας για το θέμα αυτό. Και τέλος, όσον αφορά τις ε, πολυεθνικές, δεν ξέρω τι μπορώ να προσθέσω σε αυτό. Το έχω σημειώσει, αλλά πρέπει να σας πω, δεν έχω αξιολογήσει ακριβώς αυτό το θέμα της απεικιοκρατίας που κατά κάποιον τρόπο εμφανίζεται. Κάποιες λοιπόν πολυεθνικές ε, και εδώ αναφέρομαι κυρίως σε αυτές που έχουν έδρα στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες, κάποιες ε, σημαντικές, μεγάλοι παίκτες, προφανώς και έχουν επενδύσει στις στις ευκαιρίες. το ισχύει ας πούμε για τη Microsoft, για την Google, για το Facebook. Αυτοί έχουν γίνει σημαντικοί παίκτες, ε, ε, προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις και αν δεν το έκανα, ε, ακόμα στη διάθεσή σας είμαι, είμαι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι πολλά τα ερωτήματα που σας τέθηκαν. Με αυτά ασχολούμαστε στην Επιτροπή μας και προσπαθούμε να προβάλλουμε εναλλακτικέ λύσεις. Πράγματι, είναι απογοητευτικό να διαπιστώνουμε ότι από τη μία χρονιά στην άλλη το μόνο που κάνουμε είναι να επαναλαμβάνουμε συζητήσεις. Ε, εμείς έχουμε την αίσθηση ότι τα πράγματα προχωρούν πάρα πολύ αργά. Ωστόσο, όταν κανείς δεν ξέρει πόση δουλειά έχει να, μην, έχει να γίνει ακόμα, πόση δουλειά έχει μείνει, δύσκολα ε, ξεκινάει και κινητοποιείται. Μας βοηθήσατε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στη δουλειά σας, στην έρευνα που διεξάγεται στους κόλπους της πανεπιστημιακής κοινότητας, γιατί όλα αυτά βοηθούν στην επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων, ο οποίος και μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι τα θέματα που θα συζητηθούν το απόγευμα είναι εξαιρετικά σημαντικά, όπως και η οδηγία για την άδεια μητρότητα, την οποία θα συζητήσουμε το απόγευμα. Θα συζητήσουμε επίσης για, τη ε, για την ε, συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον αγώνα έτσι ώστε να εξαλειφθεί η βία εναντίον των γυναικών. Δυστυχώς στη δική μου χώρα, στην Ισπανία, αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των γυναικών που βρήκαν το θάνατο από τα χέρια των συντρόφων τους. Ε, μιλούμε λοιπόν για την ενδοοικογενειακή βία. Πρέπει να δουλέψουμε για να πετύχουμε ισότητα στην Ευρώπη πρέπει να έχουμε επιτυχημένες στρατηγικές καταπολέμησης της βίας εναντίον των γυναικών. Θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις σήμερα το απόγευμα, όπως τις ακούσαμε σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστούμε θερμά και τις τρεις ε, ειδικού, τις τρεις εμπειρογνώμονες και καθηγήτρες για την ευελιξία σας, για την ποιότητα των παρουσιάσεών σας. Θα τα πούμε στις τρεις το απόγευμα, οπότε και θα, θα συνεχίσουμε με το εργαστήριο που έχουμε οργανώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.